οποίο επετέλεσε η κυρία εισηγήτρια Όμεν Ρόιτεν. Περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερησία διάταξή μα, που είναι οι δηλώσει του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκθεση του 2012 σε σχέση με τι πρόοδου που σημειώθηκαν όσον αφορά το Μαυροβούνιο. Και πρώτα απ' όλα θα δώσουμε τον λόγο για άλλη μια φορά στην αγαπητή Υπουργό κυρία Λουσίντα Κρέιτον, ώστε να μας εκθέσει τις απόψεις του Συμβουλίου σε σχέση με αυτό το ζήτημα για το Μαυροβούνιο. Έχετε τον λόγο κυρία Κρέιτον. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Όταν το Συμβούλιο αξιολόγησε την πρόοδο όσον αφορά τη διεύρυνση συνεδρίας 11 Δεκεμβρίου του 2012, όπως γνωρίζετε, είδε θετικά την πρόοδο στο Μαυροβούνιο όσον αφορά την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα θέματα που τονίθηκαν ήταν η ενίσχυση της λειτουργίας του Κοινοβουλίου, του δικαστικού τομέα, τη πολιτική κατά τη διαφθορά, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η προστασία των δικαιωμάτων ατόμων που ανήκουν σε μειονότητε. Ε, το Συμβούλιο επίση σημείωσε συνεχιζόμενε αλλαγέ όσον αφορά το Σύνταγμα και το δημόσιο τομέα. Ε, το Μαυροβούνιο επίση συνέχισε να εφαρμόζει ομαλά τι υποχρεώσει του παπορέων όσον αφορά τη ε, Συμφωνία Συμφωνή Σταθεροποίηση και να παίζει θετικότατο ρόλο στην περιοχή και μέσω επίκοδομητική συμμετοχής στην ανάπτυξη περιφερειακής συνεργασίας. Πολλά από αυτά τα θέματα αντικατοπτρίζονται στο ψήφισμά σας και θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερως τον εισηγητή Charles Tannock για την έκθεσή του και την θετικότητα τη συμβολή του στην προώθηση τη ενταξιακή διαδικασία για το Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο τώρα θα πρέπει να οικοδομήσει στην επιτευχθήσα πρόοδο και να παγιώσει την μεταρρυθμιστική διαδικασία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη θετικού ιστορικού στον τομέα τη εφαρμογή του κράτου του δικαίου. Βιώσιμη και διαρκής μεταρρύθμιση χρειάζεται, κυρίως όσον αφορά τη μετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και περιπτώσεις διαφθοράς και σε επίπεδο ανωτέρων στελεχών. Το Συμβούλιο καλωσόρισε την έκθεση της Ευρωπόλου όσον αφορά το θέμα του οργανωμένου εγκλήματος στο Μαυροβούνιο. Περαιτέρω προσπάθειες απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ο έλεγχος και η ανεξαρτησία του δικαστικού τομέα και να ενισχυθεί το διοικητικό δυναμικό για την εφαρμογή του κεκτημένου. Εν γέννη, οι ενταξιακέ διαπραγματεύσει ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά η Κυπριακή Προεδρία μπόρεσε να ανοίξει τα πρώτα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων με το Μαυροβούνιο, επιστήμες και έρευνα. Συγκεκριμένα, η Ιρλανδική Προεδρία κατάφερε με τη σειρά της να ανοίξει ένα δεύτερο κεφάλαιο, με τα χαράς λέω πολιτισμός και παιδεία ε, και έγινε ενταξιακή διάσκεψη που έλαβε αρχές εβδομάδας έλαβε μέρος, ε, έλαβε χώρα, συγγνώμη. Και του επόμενου μήνε θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να πετύχουν περαιτέρω πρόοδο διαπραγματεύσει και ή δυνατόν να ξεκινήσει κι άλλο ένα, να ανοίξει άλλο ένα κεφάλαιο Μαζί με τις διαπραγματεύσεις η όλη, όλος έλεγχος ε, προχωράει, πολύ καλή πρόοδος. Έλεγξε η Ευρωπαϊκή Ένωση τα κεφάλαια όσον αφορά το κάτω δικαίου, δικαστικό τομέα, θεμελιώδη δικαιώματα, δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια και εκλήθη το Μαυροβούνιο να ετοιμάσει τα απαιτούμενα σχέδια δράση που είναι τα αρχικά απαιτούμενα για αυτά τα κεφάλαια. Δεν περιμένουμε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για αυτά τα κεφάλαια κατά τη διάρκεια της ελληνική ε, Προεδρίας. Το προπαρασκευαστικό έργο που απαιτείται θα πρέπει να είναι υψής της ποιότητας και αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούμε κάποιο χρόνο όμως θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε το Μαυροβούνιο να προχωρήσει τις προσπάθειές του ταχύτερο δυνατόν. Αυτό θα επέτρεψει στο Μαυροβούνιο να αντιμετωπίσει σε αρχικά στάδια της, διεύρυ... της διαδικασίας διεύρυνσης να αντιμετωπίσει τα κεφάλαια και να δημιουργεί θετικότατο ιστορικό μεταρρυθμίσεων που είναι σημαντικότατο αυτό για το Συμβούλιο και πιστεύω και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε ότι το Μαυροβούνιο θα υποβάλει τα σχέδια δράση που απαιτούνται κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα, ώστε να μπορούν να εξεταστούν αυτά τα ζητήματα από το Συμβούλιο και σίγουρα παροτρύνουμε το Μαυροβούνιο να το κάνει αυτό. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, θα πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει να γίνουν πολλά κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Είναι πολύ σημαντικό να παραμείνει αυτή η θετική ορμή που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία, τους τελευταίους μήνες και σας διαβεβαιώ ότι η Ιρλανδική Προεδρία θα κάνει ότι μπορεί να σημειωθεί μεγαλύτερη δυνατή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα κλείνοντα να εκφράσω την εκτίμησή μου για το έργο του Κοινοβουλίου, το οποίο αναγνωρίζω και του συγητού που όλα αυτά βοηθούν την ενταξιακή διαδικασία για το Μαυροβούνιο. Πολύ στενή συνεργασία υπήρχε μεταξύ των διεθνικών οργάνων, το εκτιμώ αυτό και προσβλέπω σε συνέχιση ανταλλαγή απόψεων να λάβω υπόψη την εμπειρογνωμοσύνη σα όσο προχωράμε στι διαπραγματεύσει. Σα ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την προσοχή σα. Ε, Πολύ σα ευχαριστούμε. Τώρα θα λάβει τον λόγο εξ ονόματο τη Επιτροπή ο κύριο Φίλε, παρακαλώ. Σε ευχαριστώ, Πρόεδρε κύριε, κυρία Υπουργέ, αγαπητοί Ευρωβουλευτές. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον εισηγητή για το θέμα του Μαυροβουνίου, Charles Στάνοκ, για αυτό το σχέδιο ψηφίσματος που αντανακλά όλα τα ευρήματα της έκθεσης πρόοδου του 2012 για αυτή τη χώρα το Μαυροβούνιο συνεχίζει να καταβάλει, να σημειώνει μεγάλη πρόοδο προς, καθοδόν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίζοντας, έχοντας προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις, ανοίγοντας ναι, ένα νέο κεφάλαιο ιστορικής σημασίας στις σχέσεις αυτής της χώρας με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τω μεταξύ, περάσαμε στην ουσία της εξέτασης θεμάτων για την ε, ένταξη. Η διαδικασία εξέτασης όλων των κεφαλαίων βρίσκεται υπό εξέλιξη. Καταφέραμε προσωρινά να κλείσουμε τα κεφάλαια 25 25 επιστημών και έρευνα στο Δεκέμβριο και το κεφάλαιο 26 εκπαίδευση, παιδεία, πολιτισμικά θέματα μόλις πριν από λίγες μέρες Ξεκινήσαμε με το κράτος δικαίου και σε σχέση με τη νέα προσέγγιση εξέταση αυτών των θεμάτων και θα συνεχίσουμε αυτή την εστίαση. Και έτσι πραγματικά θα ήθελα να συγχαρώ την Ιρλανδική Προεδρία για ένα εξαιρετικό έργο που επιτελείται από πλευρά. τη. τέσσερι παρατηρήσει έχω για τι κυριότερε προκλήσει που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και έχουμε μπροστά μα στο μέλλον. Πρώτον, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην ολοκλήρωση τη ε, εξελισσόμενη ε, συνταγματική μεταρρύθμιση. Να διασφαλίσουμε λογοδοσία και διαφάνεια όσον αφορά το δικαστικό, ευθυγραμμιζόμενοι με τις συστάσεις της Επιτροπής Βενετίας, Venice Commission. Η ανάλυση αυτών των μεταρρυθμίσεων θα έχει κέρια σημασία για τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, κάποια πρόοδο σημειώθηκε στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Όμως ο αριθμός των περιπτώσεων υπό των διώξεων και των κατα... της... Ε, του ποσοστού ε, κατά καταδικών που έχουν ε, επιτευχθεί είναι χαμηλό επιπλέον πλήρη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ε, σε σχέση με αυτόν τον τομέα είναι σημαντικό στοιχείο απαραίτητο στοιχείο για το Μαυροβούνιο για να μπορέσει να ολοκληρώσει και να συνεχίσει την ευρωπαϊκή πορεία ολοκλήρωσης. Η προστασία και η ελευθερία των μέσων ενημέρωση και του τύπου πρέπει να διασφαλιστεί. Και έτσι οι αρχές του Μαυροβουνίου σε όλα τα επίπεδα πρέπει να ενθαρρυνθούν, να αυξήσουν τις προσπάθειές τους, να υποβάλουν και πολύ νωρί να μπορούν να ε, εξηχνιάζονται τέτοιε περιπτώσει Τέταρτον, περαιτέρω προσπάθειες απαιτούνται για να βελτιωθεί η κατάσταση των συγκάλων και της ε, ε, περίπτωσης ε, των μειονοτήτων διασφαλίζοντας τα πολιτικά δικαιώματά τους, μειονοτικά δικαιώματά τους και κοινωνικά δικαιώματά τους ο διάλογός μας με το Μαυροβούνιο σε σχέση με αυτές τις ε, προκλήσεις που πρέπει ακόμα να αντιμετωπιστούν θα καθορίσουν το ρυθμό των διαπραγματεύσεων και την ταχύτητά τους. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, μια σύντομη παρατήρηση να κάνω σε σχέση με τις πρόσφατες προεδρικές εκλογές ε, που βρίσκονται υπό αμφισβήτηση ως ε, διεργασία. Είναι μια χώρα το Μαυροβούνιο που διαπραγματεύεται την ιδιότητα κράτους μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα παράπονα και οι προσφυγές πρέπει με ταχύ τρόπο να εξηχνιάζονται και να διευθετούνται το αποτέλεσμα των εκλογών πρέπει να υπό αυτό το πρίσμα να αντιμετωπιστεί. Ευελπιστώ ότι οι ηγέτες του Μαυροβουνίου θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να υπάρξει ένα αναγκαίο πλαίσιο ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία από κομματικά συμφέροντα. Ευχαριστώ. Μισά... Πρόεδρος, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα δώσουμε τώρα τον λόγο στη συνέχεια σε αγορητές που θα παρέμβουν εξ ονόματος των κοινοβουλευτικών ομάδων τους. Πρώτον, πρώτος ο δόκτωρ κύριος που θεωρώ, μια και είναι και εισηγητή κιόλα για το θέμα του Μαυροβουνίου, έχει προτεραιότητα, είναι πρώτο που θα λάβει τον λόγο. Έχετε τον λόγο παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, είναι τιμή μου να είμαι εισηγητή για το Μαυροβούνιο σε αυτό το κοινοβούλιο. Είναι μια μικρή και όμορφη χώρα που μπορεί να συνεισφέρει στην ε, παγκόσμια σκηνή και στην ε, παγκόσμια ιστορία ε, και μέσω τη ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στα κεφάλαια ε, για ε, ε, την εκπαίδευση και όλα τα κεφάλαια που έχουν εξεταστεί μέχρι τώρα βλέπουμε τα βήματα που έχουν γίνει προς την ένταξη και είναι και ένα υπόδειγμα για τις υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Θα μπορούσε λοιπόν να σκεφτεί κάθε χώρα ότι μπορεί να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Δεν μπορούμε βέβαια να αγνοήσουμε κάποια προβλήματα στη διαδικασία ένταξης του Μαυροβουνίου. Έχω κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματο και την εκπαίδευση των δικαστών όσον αφορά την καθυστέρηση των δικαστικών διαδικασιών. Επίση, θα πρέπει ε, να αντιμετωπιστεί η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα. Επίση, θα μπορούσε να θεσπιστεί ένα κώδικα διοντολογία για του ε, εκλεγέντε πολιτικού. και θα πρέπει το Κοινοβούλιο στο Μαυροβούνιο και οι ε, μη κυβερνητικέ οργανώσει και η κοινωνία των πολιτών να συμμετάσχουν περισσότερο ενεργά στη διαδικασία ένταξης Όλες οι επιθέσεις κατά των δημοσιογράφων θα πρέπει να ελεγχθούν, ε, να διερευνηθούν και να ε, καταδικαστούν. Ε, χαιρετίζω την εκλογή του νέου Προέδρου του Μαυροβουνίου. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες καταγγελίες σχετικά με τα αποτελέσματα, αλλά δεν έχω δει στοιχεία που να δείχνουν ότι έγιναν εκλογές που δεν ήταν ελεύθερες και δημοκρατικές. Ζητώ λοιπόν από όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις να συνεργαστούν στο πνεύμα του δημοκρατικού διαλόγου ε, ούτως ώστε να συνεργαστούν και προς την ένταξη της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η μικρή και όμορφη χώρα όπως την αποκαλώ πάντα μπορεί να έχει ε, τις ε, θεμητές προσδοκίες της για ένταξη στην οικογένεια των Ευρωπαϊκών κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Τάνοκ. Ευχαριστούμε κύριε Τάνοκ. Τώρα θα λάβει τον λόγο για το ΕΛΚ για δυόμιση λεπτά η κυρία Ιμπρισάγκητς παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να αναφερθώ και να πω ότι όταν επρόκειτο να ληφθεί η απόφαση όσον αφορά το Μαυροβούνιο και τις διαπραγματεύσεις συζήτησα με αρκετούς ε, που θα έπρεπε να λάβουν αυτή την απόφαση και τότε κάποιοι από τους εταίρους είπαν ότι δεν ήταν έτοιμο το Μαυροβούνιο με τις μεταρρυθμίσεις. Υπήρχαν λέει προβλήματα με το οργανωμένο έγκλημα. Η, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος δεν ήταν επαρκώς πλήρης και δεν ανταποκρινόταν στις προδιαγραφές και προσδοκίες μας και πολλά έπρεπε να γίνουν ακόμα. Τα δικά μου επιχειρήματα για να αντιμετωπίσω αυτές τις θέσεις ήταν λέγοντας ακριβώς για αυτούς τους λόγους πρέπει να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Μαυροβούνιο. Διότι θα είναι μια ευκαιρία να ασκήσουμε μοχλικά πίεση, να μοχλεύσουμε τα πράγματα ώστε να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσει. Και αυτό είναι ακριβώς εκείνο το οποίο συνέβη. Και μετά από εσά, Επίτροπε, και σε σχέση με την ε, δική σας ε, φάνταστη προσέγγιση σε σχέση με τι διαπραγματεύσει με τα κεφάλαια 22 και 23 ήταν πραγματικά ιδιοφυή αυτή η έμπνευση κατά τη διάρκεια τη εντολή σα. Αυτό είναι κάτι που απόφαση θα το θυμούμε πάντα. Είναι το καλύτερο το οποίο μπορούσε να συμβεί και συνέβη για αυτή τη χώρα και για όλες τις χώρες αυτής της περιοχής ε, για τις διαπραγματεύσεις. Ε. Και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει αρκετός χρόνος στη διάθεσή μας να υπάρξουν οι βελτιώσεις που απαιτούνται ακριβώς σε αυτούς τους τομείς. Όσον αφορά τώρα τις προεδρικές εκλογές, θα ήθελα να δώσω συνέχεια στα σχόλια που αναφέρθηκαν από τον κύριο Τάνο πιο πριν. Ο ΑΣΕ ε, συνέταξε μια έκθεση και σύμφωνα με αυτή την έκθεση ήταν ελεύθερες και δίκαιες οι εκλογές. Και δεν είδαμε καμιά άλλη επίσημη έκθεση που να λέει κάτι το διαφορετικό ή να αντιβαίνει αυτές τις ε, πιστώσεις. Θέλουμε λοιπόν έτσι την επίσημη αυτή έκβαση των εκλογών να την αναγνωρίσουμε. Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά βιβαιότητα για αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να έχουμε μια θετική προσέγγιση όσον αφορά τα θεσμικά όργανα και μέσα στα θεσμικά όργανα πρέπει να επιτευχθεί μια συμφωνία και πρόοδος. Είναι ένας τρόπος να καταδειχθεί ότι είναι βιώσιμη κατάσταση και είναι ικανή αυτή η χώρα να αντιμετωπίσει το μέλλον στην πορεία της. Αυτό θα είναι κέριος παράγοντας για την λήψη απόφασης από πλευράς μας για αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστούμε κυρία Εμπρισάγεβιτς. Για τους σοσιαλιστές, δημοκράτες και σοσιαλιστές, δυόμιση λεπτά ο κύριος Ρούτσεκ παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι, μετά την 1η Ιουλίου, μετά την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Μαροβούνιο θα είναι στην πρώτη γραμμή από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που κινούνται προς την ένταξη και το Μαυροβούνιο μπορεί να είναι ένα σαφές παράδειγμα πρόοδου στην περιοχή. Ένα παράδειγμα το ότι μπορεί να επιτευχθεί κάτι αν η χώρα πραγματικά επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στις μεταρρυθμίσεις παρότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο, πιστεύω ότι το Μαυροβούνιο έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά του. Θα πρέπει να επιταχύνει τις προσπάθειες ε, για τη δημιουργία αποτελεσματικού και αμερόληπτου δικαστικού σώματος ε, και να διευρύνει την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ακόμη θα πρέπει να αποπολιτικοποιήσει και να κάνει αξιοκρατική τη δημόσια διοίκηση θα πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι θεσμοί για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων σε όλους τους άλλους τομείς επίσης. Υπάρχουν ανησυχίες ε, για τον τομέα της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, την δυνατότητα των δημοσιογράφων να ασκούν κριτική κατά των τον εξουσία. Και αυτό είναι μια θεμελιώδης αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, διότι τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης που ασκούν κριτική δίνουν ε, τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται μια αποτελεσματική κυβέρνηση. Τέλος, πιστεύω ότι το Μαυροβούνιο θα πρέπει να επικεντρώσει το ενδιαφέρον ενδιαφέρον του στι μεταρρυθμίσει για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και αυτό θα πρέπει να είναι μια βασική προσπάθεια για όλα τα πολιτικά κόμματα. Όταν γίνονται οι εκλογέ, μετά τι εκλογέ δεν θα πρέπει να αποπροσανατολίζονται από άλλα τοπικά ζητήματα ε, τη χώρα. Η ομάδα μας υποστηρίζει τη διαδικασία διεύρυνσης ε, εφόσον το Μαυροβούνιο ε, τηρεί αυτή την ταχεία πορεία προς την ένταξη. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρόντσεκ. Για τους ε, δημοκράτες και φιλελεύθερους για δύο λεπτά ο κύριος Βάιγκλ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόεδρε, επίτροπε, κυρία Υπουργέ, δύο μέρες πριν μόλις. Όπως προηγούμενα προανέφερε η κυρία Υπουργό, η διάσκεψη για την ένταξη του Μαυροβουνίου ε, έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες και εκεί το δεύτερο κεφάλαιο άνοιξε και είχαμε και το κεφάλαιο 26 για τον πολιτισμό και τα συναφή θέματα. Όλα αυτά έχουν σημαντική συμβολική σημασία. Δίνουν στους νέους Μαυροβούνιους δυνατότητα να συμμετέχουν σε θελκτικά προγράμματα όπως το Erasmus Mundus και άλλα σημαντικά προγράμματα. Ένα παράθυρο που ανοίγει για αυτούς τους νέους στον κόσμο και για τη σημασία και σπουδαιότητα για το πώς έχει προπαρασκευαστεί το Μαυροβούνιο για αυτές τις, προ... Ε, για αυτές τις διαπραγματεύσεις υπό την Ιρλανδική Προεδρία το η πρόταση ψηφί ψηφίσματος του συναδέλφου ε, Τάνοκ αναφέρει και άλλες πρόοδους ε, του Μαυροβουνίου που έχουν ε, σπουδαιότητα, έχουν τη σημασία τους και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται λόγος και για άλλους τομείς όπου έχει πολλά να πράξει ακόμα το Μαυροβούνιο. Μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα. ε, συνεχίζοντα τη συστηματική μάχη κατά της διαφθοράς, δημιουργώντα μια σύγχρονη κυβερνητική δομή και κυβερνητικέ αρχέ. Οι πρόσφατε προεδρικέ εκλογές που σύμφωνα με τους παρατηρητές διεξήχθησαν σύμφωνα με δημοκρατικές αρχές δείχνουν τις διαχωριστικές γραμμές που υφίστανται στην ίδια την κοινωνία του Μαυροβουνίου όσον αφορά την θρησκεία και την εθνοτική ε, καταγωγή. Και όλα αυτά ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα μπορέσουν να οδηγήσουν στο να επιτευχθούν συμβιβασμοί και να υπάρξει προσέγγιση και άλλων τομέων και να μπορέσει καμιά φορά να μπορέσουν επίμαχα θέματα να κλείσουν. Ε, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα, όμως για το Μαυροβούνιο πρέπει να τονίσουμε τη σπουδαιότητα αυτής της ψηφοφορίας. Έχει μεγάλο ρόλο για τη σταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής το Μαυροβούνιο. Με χαρά θα παρακολουθήσουμε την πρόοδο του Μαυροβουνίου τους επόμενους, κατά την επόμενη περίοδο. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια εξ ονόματος της Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για 1,5 λεπτό κυρία Λούνατσεκ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και Επίτροπε. Κύριε Υπουργέ, το Μαυροβούνι είναι μια όμορφη χώρα όπως ήδη ελέγχθη. Έχει όμορφα τοπία, ωραίους ανθρώπους, ωραίες παραδόσεις. Ε, η πολυμορφία τη χώρας είναι σημαντική και πρέπει να προσπαθήσουμε να την διατηρήσουμε. Και θα πρέπει και τα οικολογικά μελήματα να αντικατοπτρίζονται στο Σύνταγμα. Και θα πρέπει να μας απασχολήσουν και θέματα όπως ανανεώσιμες ενέργειες, αλλά και ο τουρισμός θα πρέπει να διατηρεί το φυσικό κάλο της χώρα Θα πρέπει λοιπόν ε, να διατηρήσει την πολυμορφία του και δημοκρατία και το κράτος δικαίου θα πρέπει να λειτουργούν υπέρ των, των συμφερόντων των πολιτών. Χαιρετίζουμε το ότι το Μαυροβούνιο είναι η επόμενη χώρα που διαπραγματεύεται την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό ότι η Κροατία θα γίνει ε, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι σημαντικό το ότι έχουμε την επόμενη χώρα που παίρνει σειρά και θα έρθουν και άλλες χώρες. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες ε, κριτικές τις οποίε θα ήθελα να εκφράσω, Ιδίω για δύο σημεία τα οποία ανησυχούν και εμένα και την ομάδα μου. Το ένα είναι η ανεξαρτησία και ελευθερία των μέσων ενημέρωση. Και θα ήθελα να δείξω ένα συγκεκριμένο θέμα, μια συγκεκριμένη υπόθεση δύο δημοσιογράφων, κατά των οποίων υπάρχει μια μήνυση από την αδελφή του Πρωθυπουργού για αυτά τα οποία έγραψαν σχετικά με την εμπλοκή τη στην ιδιωτικοποίηση των τηλεπικοινωνιών. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει λοιπόν να διερευνηθεί διότι δημιουργούνται ανησυχίε ε, από τέτοια γεγονότα. Και το δεύτερο είναι οι πρόσφατες προεδρικές εκλογές έχουν αμφισβητηθεί από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από πολλέ μη κυβερνητικέ οργανώσει. Και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το Μαυροβούνιο να δείξει το δημοκρατικό του χαρακτήρα, να, δείξει, να γίνει λοιπόν πλήρη διερεύνηση όλων αυτών των καταγγελιών, ώστε να μην υπάρχουν πολιτικά συμφέροντα. Και ελπίζω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι για την τροπολογία αυτή θα με υποστηρίξετε αύριο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, τώρα θα λάβει τον λόγο εξ ονόματος της Ενωτικής Αριστεράς και Πράσινης Βόρειας Αριστεράς για ένα, μισή λεπτό. Ο κύριος Χουντής παρακαλώ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι η υπόθεση του Μαυροβουνίου είναι από τις πιο εύκολες περιπτώσεις διεύρυνσης από τις χώρες των Βαλκανίων. Όμως υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά αν όλη αυτή η διαδικασία αποβλέπει στην ευημερία των πολιτών πράγματι το μαυροβούνιο πληρεί αρκετά από τα ενταξιακά κριτήρια πράγματι πρέπει να λυθούν έτσι κι αλλιώ προβλήματα που καταγράφει η έκθεση όμω δεν βελτιώνεται η κατάσταση του λαού του μαυροβουνίου και η καθημερινότητα. η ανεργία αυξάνεται κατά επίσημα στοιχεία συνεχώ. υπάρχει ανεργία ανέχεια υπάρχει φτώχεια και υπάρχουν τέτοια κοινωνικά προβλήματα. τα μέτρα που λαμβάνονται υποτίθεται για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα είναι ανεξέλεγκτη ανεξέλεκτες ξένες επενδύσεις που έχουν μεταβάλει το μαυροβούνιο ως μια χώρα από τις πιο σημαντικές που ξεπλένεται μαύρο χρήμα. δεύτερον επενδύσεις και ιδιωτικοποίησεις που σημαίνει ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου. τρίτον επενδύσεις καταστροφικές για το περιβάλλον που είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για ήπια τουριστική ανάπτυξη. αγαπητοί συνάδελφοι κύριε επίτροπε κύριε κυρία υπουργέ τα οικονομικά κριτήρια που προτείνονται για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση και που ζητιούνται είναι στην ίδια κατεύθυνση. πρέπει να ξέρουμε ότι στους λαούς των βαλκανίων που αυτή η πορεία έδινε κάποιες ελπίδες έχει διαψευστεί λόγω της οικονομικής κρίσης της ευρωπαϊκής ένωσης. δεν το βλέπουν ως ελκυστικό πια αυτό το όραμα. επομένως ε, αγαπητοί φίλοι αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε υπουργέ και κύριε επίτροπε υπάρχει πάρα πολύ σημαντικό θέμα το τι ζητάμε και προς τα ποια κατεύθυνση ζητούμε να λυθούν και αυτά τα προβλήματα όχι μόνο αυτά που αναφέρονται και για τα οποία συμφωνώ πολύ Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε κύριε Χούντι. Περνάμε στου άλλου αγορητέ. Δύο λεπτά ο κύριο Κούκαν. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, κυρία Υπουργέ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Τσάρλ Στάνοκ για την σύνταξη αυτής της ε, ισόρροπης ε, έκθεσης και σε σχέση με την διαδικασία ολοκλήρωσης στα Βαλκάνια που είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε. Η έναρξη των διαπραγματεύσεων ενισχύει τις μεταρρυθμίσεις σε αυτή τη χώρα, στο Μαυροβούνιο. Και γι' αυτό θέλω να απευθύνω έκκληση να συνεχιστεί από το Μαυροβούνιο η προσπάθεια των μεταρρυθμίσεων. Το έργο αυτό το οποίο βρίσκεται μπροστά τους και πρέπει να αντιμετωπιστεί αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Θα είναι αναγκαίο να υιοθετηθούν και να εγκριθούν σημαντικά μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνεια. Τη της χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων, της ε, πολιτικής ε, ζωής ε, και πολιτικών εκστρατιών για να μπορέσει να βελτιωθεί η καταπολέμηση της διαφθοράς. Ένα σημαντικό στοιχείο για τα οικονομικά κριτήρια τα οποία έχει επιτύχει αυτή η χώρα πρέπει να οδηγήσει στην παγίωση, στην έδραση αυτών των στοιχείων, να δημιουργηθεί ένα σταθερό, αξιόπιστο δημοκρατικό σύστημα. Πρέπει να συνεχιστεί το έργο το οποίο ανελήφθη και πρέπει αυτά τα οποία είδαμε σε σχέση με τις ε, προεδρικές εκλογές να πούμε ότι μας υπενθυμίζουν πόσο ευαίσθητα απομένουν και εξακολουθούν να είναι όλα αυτά τα ζητήματα. Αφενός πρέπει να αποσαφινιστούν όλα τα θέματα που εκκρεμούν όσον αφορά αυτές τις ε, προεδρικές εκλογές και πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι η κοινοβουλευτική υπονόμευση δεν είναι η σωστή πορεία. Επίσης ε, πρέπει να αναφέρουμε ότι η διαδικασία των διαπραγματεύσεων ένταξη του Μαυροβουνίου στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα προς τις άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παρακολουθήσει λοιπόν εκ του σύνεγγυς όλα αυτά και να υπενθυμίσει στις χώρες αυτές ότι πρέπει να αρθούν στο ύψος των κριτηρίων της Κοπεχάγης για να συνεχίσουν την πρόεδρο. Και τώρα για δυόμιση λεπτά θα λάβει τον λόγο ο κύριος Ζάλα. Αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ συχνά Ακούω ότι τα κριτήρια για την εισδοχή, για την ένταξη του Μαυροβουνίου είναι κάτι απλό. Η ιδέα ότι ο δρόμος του Μαυροβουνίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εύκολος. Αλλά πόρο απέχει από την αλήθεια αυτή η εντύπωση και πρέπει να θυμόμαστε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι μετά την ένταξη της Κροατίας η αδίποτε ενταξιακή διαδικασία που θα ακολουθήσει θα δυσχεραίνει. Οι κανόνες θα είναι πιο αυστηροί και το άνοιγμα, η ανοιχτή θέση των κρατών μελών για τη διεύρυνση θα κλείνει συνέχεια. Συμφωνώ, τον Τζαλτ Στάνοκ, τον εισηγητή του Μαυροβούνιο, πρέπει να συνεχίσει τι μεταρρυθμίσει του, κυρίω του δικαστικού τομέα και στον τομέα καταπολέμηση διαφθορά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν τα μέσα ενημέρωση. Όλα αυτά πρέπει να απειληθούν. Το Μαυροβούνιο δεν μπορεί να έχει πολιτικέ κρίσει. Ακολουθεί το σωστό δρόμο η χώρα και ηγείται στην ε, περιοχή, όπως ήδη αναφέρθηκε και από άλλους ε, αγορητές. Όμως το Μαυροβούνιο δεν μπορεί να υποτιμά την ενταξιακή διαδικασία. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Σας ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα στον γύρο Catch Για ένα λεπτό. Ο κύριος Ζένκε, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω Σα ευχαριστήσω που μα δίνετε τη δυνατότητα να συζητήσουμε, διότι η δυνατότητα ένταξη του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ειδωθεί από διάφορε οπτικές γωνίες. Δηλαδή μπορεί να το δει κανεί από την νομική σκοπιά ε, και από την ε, πολιτική σκοπιά. Αν το δει κανεί από την νομική σκοπιά, ευτυχώ μιλάμε για μια χώρα που έκανε σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του νομικού συστήματο, την καταπολέμηση τη διαφθοράς και τα δικαστήρια είναι ανεξάρτητα και υπάρχει ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Όμως υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο, μια δεύτερη οπτική γωνία η οποία πιστεύω ότι είναι σημαντική στην περίπτωση της συγκεκριμένης χώρας. Προφανώς θα πρέπει να εγγυηθούμε την ασφάλεια στην Ευρώπη και αυτό που είναι σημαντικό στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι το Μαυροβούνιο προφανώς θα πρέπει να βελτιώσει την κατάσταση και να στεθεροποιήσει την κατάσταση στα Βαλκάνια. Μιλάμε για μια περιοχή με πάρα πολύ δύσκολη, δύσκολο ιστορικό και πάντα υπήρχαν συγκρούσεις και πόλεμοι στην περιοχή. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ζένκε. Τώρα θα λάβει τον λόγο ο κύριος Μέλτσερ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε η αντιμετώπιση μιας εκλογικής διαδικασίας δίνει κάποια συμπεράσματα για την δημοκρατική οριμότητα μιας χώρας. Όσον αφορά όμως λαθροθυρίες ε, και ε, κάποιες ε, τέτοιες, κάποιους τέτοιους ελιγμούς δεν είναι υπέρ της, του Μαυροβουνίου για την Ποντγκόριτσα αληθεύει ότι είχε συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία και είχε χάσει κατά κάποιο τρόπο τους στόχους ενώπιον της η χώρα αυτή. Είχε πει ένα ολόκληρο έτος αποκλειστικά λογική αντιπαράθεση. Δεν πρέπει όμω οι μεταρρυθμίσει να παραμεληθούν περισσότερο. Επιτέλου ήρθε η χρονική στιγμή να ασκηθεί η επιρροή ώστε σε σχέση με το δικαστικό, την καταπολέμηση τη διαφθορά, την διασφαλίση τη ελευθερία του τύπου και των μέσων να σημειωθούν πρόοδοι. Να αρθεί στο ύψο των περιστάσεων το Μαυροβούνιο και να προσεγγίσει τι προδιαγραφέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο έτσι μπορεί να έχει μια ευρωπαϊκή προοπτική. Έτσι λοιπόν η προσχώρηση, η ένταξη τη Κροατία μπορεί να αποτελεί ένα ορόσημο για τι ε, χώρε τη πρώην Ιουγκοσλαβίας που μπορούν να ακολουθήσουν την ίδια πορεία μελλοντικά. Σα ευχαριστούμε κύριε Μπέλτσερ, λέει ο Πρόεδρο Και τώρα για ένα λεπτό ο κύριο Κατσίν, παρακαλώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για ε, την έκθεση αυτή και συγχαίρω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κλείσιμο ε, των κεφαλαίων αυτών. Δείχνει ότι ήταν καλή οργάνωση και επιτυχής η εργασία τους όσον αφορά τη χώρα αυτή ε, Ποια είναι τα θεσμικά όργανα στα οποία υπάρχουν εμπόδια. Δεν είναι το Κοινοβούλιο και ο Πρωθυπουργό. Ε, και αυτό το μήνα θα γίνει η συνάντηση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μαυροβουνίου και δεν θα πρέπει ε, να ε, μπλοκάρει κανεί αυτή την συνέλευση. Γιατί δεν μιλάμε για την Αλβανία. Μιλάμε για μια χώρα που βρίσκεται υπό μεταρρύθμιση. Δεν θα πρέπει λοιπόν κανεί να θέσει εμπόδια στην συνέλευση δεν είναι σωστός τρόπος για την προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει τα προβλήματα να επιλύονται με θεσμικό τρόπο και σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία θα πρέπει το Κοινοβούλιο να παίζει το... Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κατσίν. Τώρα θα λάβει τον λόγο ο Επίτροπος κύριος Φίλε, παρακαλώ. Commissioner, Επίτροπε, έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, Υπουργέ, αξιότιμα μέλη. Θα ήθελα να ολοκληρώσω τα σχόλιά μου επαναλαμβάνοντας τα συγχαρητήριά μου προς τον εισηγητή, τον Τσουαλ Τάνοκ. Πολύ υψηλή ποιότητα της έκθεσής του. Παραδέχτηκε, αναγνώρισε την επιτευθύσα πρόοδο και έτσι στέλνουμε ένα ισορροπημένο μήνυμα που θα πρέπει να ενθαρρύνει το Μαυροβούνιο να αυξήσει τις μεταρρυθμίσεις καθοδόν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τι συνεδριάσει εξέταση και ανείχνευση τη προόδου την περασμένη άνοιξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη προετοίμασε την έκθεση αυτή τη διήθηση για τι διαπραγματεύσει των διαφόρων κεφαλαίων για το δικαστικό τομέα και θεμελιώδη δικαιώματα, δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια, 23 και 24. Και το Μαυροβούνιο προσεκλήθη από το Συμβούλιο το Δεκέμβριο να ετοιμάσει το σχέδιο δράσης που απαιτούνται και να αρχίσει η βαθμολόγηση και για τα δύο κεφάλαια και ο έλεγχος. Η πρόοδος του Μαυροβουνίου αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις στους συγκεκριμένους ε, τομείς, στα συγκεκριμένα κεφάλαια που αφορούν το κράτος δικαίου, ε, όλα αυτά θα επηρεάσουν άμεσα την πορεία των διαπραγματεύσεων, το ρυθμό. Οι ενταξιακέ διαπραγματεύσει θα είναι πολύ απαιτητική διαδικασία για το Μαυροβούνιο, αλλά πιστεύω ότι με την κοινή μα υποστήριξη και με την ισχυρή αφοσίωση ε, του Μαυροβουνίου στην πορεία του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει η χώρα αυτή να εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος των πολιτών του και θα θέσει ένα ε, θετικό παράδειγμα στα Δυτικά Βαλκάνια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε και τώρα δίνουμε το λόγο στην κυρία Κρέιτον εκ μέρου του Συμβουλίου. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ξεκινώντας, θα ήθελα να υποστηρίξω τις θέσεις του κυρίου Τάνοκ για το Μαυροβούνιο, ότι είναι μια μικρή και όμορφη χώρα. Όντως είναι μια πανέμορφη χώρα. Και συμφωνώ ότι είναι μια χώρα που έχει πάρα πολλά να συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια και προσβλέπω σε αυτή τη συνεισφορά του Μαυροβουνίου εν ευθέτω χρόνο. Η ένταξη είναι βέβαια ένα πολύπλοκο ε, θέμα και συχνά είναι και μια διαδικασία που έχει πολλές απογοητεύσεις. Αναφίβολα, οι χώρες ε, που υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, λαμβάνονται υπόψη όχι ε, μόνο με βάση το κοινωτικό κεκτημένο, αλλά σε μεγάλο βαθμό. Αυτό δεν είναι κάτι που θα πρέπει να φοβούνται οι χώρες αυτές. Είναι μια θετική ευκαιρία και για την υποψήφια χώρα, για το Μαυροβούνιο στη συγκεκριμένη περίπτωση, και για τις υφιστάμενες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλαίσιο διαπραγμάτευση για το Μαυροβούνιο ε, όντως ε, θέτει σε λειτουργία αυτή την προσέγγιση σχετικά με πρόοδο σε θέματα κράτους δικαίου για τα κεφάλαια ε, που συνδέουν την πρόοδο με τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη και νομίζω ότι το Μαυροβούνιο πηγαίνει αρκετά καλά. Τα κεφάλαια που αφορούν το κράτος δικαίου τα αντιμετωπίζουμε στην αρχική διαδικασία των διαπραγματεύσεων για να υπάρξει επαρκής χρόνος για να δημιουργηθούν οι απαραίτητοι θεσμοί και για να, υπάρξει, να υπάρξουν τα κατάλληλα βήματα πριν από το κλείσιμο των διαπραγματεύσεων. Και αυτό ε, προσθέτει αξιοπιστία στη διαδικασία διεύρυνσης και είναι κάτι το οποίο θεωρώ ιδιαίτερα θετικό. Η επιτυχία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το ίδιο το Μαυροβούνιο, αλλά ε, είμαστε πρόθυμοι για να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Ε, προσβλέπουμε λοιπόν στη στενή συνεργασία μαζί σας με τους φίλους μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας όχι μόνο όσον αφορά ε, την ενταξιακή διαδικασία για το Μαυροβούνιο αλλά και για τις άλλες υποψήφιες χώρες και θα συνεχίσουμε ε, σε αυτό το πνεύμα συνεργασίας και μετά την Ιρλανδική Προεδρία. Βασιζόμαστε λοιπόν στην υποστήριξή σα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βασιζόμαστε στην εταιρική σχέση μαζί σα για να διατηρήσουμε και την υποστήριξη των πολιτών μα σε μια κοινή προσπάθεια που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική όπω σα είπα ήδη. Σα ευχαριστώ λοιπόν για άλλη μια φορά για την εξαιρετική συζήτηση ε, που έγινε. σα ευχαριστώ για το πνεύμα συνεργασία ε, για το θετικό πνεύμα που υπάρχει στην Ολομέλεια και σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κρέιτον. Έχουμε το ψήφισμα για αυτό το θέμα τώρα. Θα το ψηφίσουμε αύριο στις 11.30. Και προχωρούμε.